it was on already, so everybody heard what we are preparing. Okay. Hi. So, uh, well, I, uh, dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, μου συνέστησα να χρησιμοποιώ και το σφυράκι και αυτό θα κάνω. Θα ήθελα να αρχίσουμε στη σημερινή μας συνεδρίαση. Νομίζω πρώτα απ' όλα θα έπρεπε να, να σας καλωσορίσω όλους μετά τις διακοπές. Σίγουρα παραμείνατε δραστήριοι και εσείς και οι συναδελφοί σας, ε, διότι συνέβησαν πολλά τις τελευταίες εβδομάδες. Στη επηρέασαν την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα τα συζητήσουμε. Έχετε την, το σχέδιο ημερήσια διάταξη. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, θα πρότεινα να εγκρίνουμε το σχέδιο ημερήσια διάταξη. Ωραία, ευχαριστώ. Α περάσουμε στο δεύτερο σημείο, έκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων των 15 και 16 Ιουνίου 2015 και 29 Ιουνίου 2015. θα θεωρηθούν εγκεκριμένα εάν δεν υποβάλλεται σχόλια, ενστάσεις μέχρι το πέρα συνεδρίαση, ως συνήθω. Σημείο 3. Ανακοινώσει του Προέδρου. Αναμεταδίδεται η συνεδρίαση ως ήθιστε και έχουμε και τη διερμηνία. Θα ήθελα να μιλάτε με ε, όχι υπερβολικά γρήγορο ρυθμό για να διευκολύνετε το έργο των διερμηνείων. Εάν υπάρχουν ερωτήσεις μπορείτε σε σχέση με αυτά που σας έχουμε ε, διανύμει να τις απευθύνετε στη γραμματεία. Ε, για την Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου με το Βιετνάμ, 1η Αυγούστου ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι επί της αρχής έχουμε καταλήξει συμφωνία με το Βιετνάμ μετά από 2,5 χρόνια έντονων διαπραγματεύσεων. Σε αυτή την ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε ότι επήλθε συμφωνία για όλα τα ουσιαστικά ζητήματα και είναι αμοιβαίως επωφελής και ισόρροπη η συμφωνία. Και συμπλήρωσε ότι οι διαπραγματευτικές ομάδες θα συνεχίσουν τώρα τη διαδικασία, θα ρυθμίσουν κάποια εκκριμή ζητήματα και θα καταλήξουν σε ένα οριστικό ε, νομικό κείμενο το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από πλευρά ε, τη Επιτροπής θεωρώ ότι αυτά είναι πολύ καλά νέα και θα ήθελα να συγχαρώ επί τη ευκαιρία τη διαπραγματευτική ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως ξέρετε, ήταν ύψιστη προτεραιότητα για μας η διαπραγμάτευση της συμφωνίας με το Βιετνάμ και στο Ανόη και στο Χωσιμίχ πήγαμε εξάλλου τον Απρίλιο με μεγάλη αντιπροσωπή από πλευρά μα, ε, εν και της μελλοντική συμφωνία. Ε, συναντήκαμε τον Πρωθυπουργό του Βιετνάμ για να αναφέρουμε ποιε είναι οι δικέ μα προτεραιότητε εδώ στην Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου και στην Επιτροπή Παρακολούθηση, όπου προεδρεύει ο κύριο Σαχράου, που είναι ο μόνιμο ηγητή μα. Παρακολούθησε τη διαδικασία και θα συνεχίσει να παρακολουθεί το πέρα τη διαδικασία, ούτω ώστε να είναι ε, ολοκληρωμένη, ισόρροπη και αμοιβέ υποφελή η συμφωνία. Επίσης υπάρχει και η συμφωνία για τα περιβαλλοντικά αγαθά και έγινε ο 8ος ο οποίος ολοκληρώθηκε στις 31 Ιουλίου το, τη Γενέ, στη Γενέβη και έχουμε λάβει από πλευρά της Γραμματείας το κείμενο της Διπουργικής Συμφωνίας. Στο σχέδιο βλέπουμε διάφορα κεφάλαια όπου καλύπτονται ζητήματα όπως θεσμικές ρυθμίσεις, ζητήματα χρονισμού και θα επεξεργαστεί θα επεξεργαστούν και τον κατάλογο των αγαθών το Σεπτέμβριο από τις 16 μέχρι τις 22 στον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων δηλαδή ε, στη συνέχεια η διάσκεψη των πρέσβων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα συναντηθούν μαζί μας στις 2 Σεπτεμβρίου οι μόνιμη αντιπροσωπείες ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διοργανώνουν τη διάσκεψη, η οποία θα γίνει σε δύο μέρη. Στην Ολομέλεια ε, περιορίζεται η συμμετοχή των επιτροπών στου προέδρους και του συντονιστές. Ακολουθούν διάφορε συνεδριάσει ε, όπου θα παρευρεθούν και οι μόνιμοι εισηγητέ των επιτροπών μα, Ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Στι εξωτερικέ δράσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσουν ο τίτλο και ο στόχο αυτή τη διάσκεψη. Στη συνέχεια, η Φεντερίκα Μογκερίνη, αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απήντησε στην επιστολή του Προέδρου Λάγκη και του Πρόεδρου Μπρόκ ε, εν ώψη και τη συνόδου με την Ιαπωνία η απήντησε η, στην επιστολή λοιπόν η Φεντερίκα Μοκερίνη, Επίσης, η κυρία Αρμόδια Επίτροπος Μάλμστρομ είχε αποστείλει αντίστοιχη επιστολή και απήντησε η κυρία Μογκερίνη ότι υπάρχει σε μεγάλο βαθμό σύγκληση σε σχέση με τον προσανατολισμό για τη στρατηγική εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας. Επίσης, υπάρχει μια ε, σειρά από βασικά ζητήματα ε, στρατηγική σημασία που έχει διετονίσει η Επιτροπή μα εν ώψη τη διάσκεψη και αυτά απαριθμούνται μέσα στην επιστολή. Αυτά έχω να αναφέρω και ο κύριο Μπέγκε, όχι ο κύριος Λάγκη, ο κύριος Μπέγκε που είναι εισηγητής ε, για τον προπολογισμό 2016 θα έρθει. Έχουμε ήδη συζητήσει το ζήτημα, έχουμε την γνωμοδότηση τη Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου Σίγουρα θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι η ενόψη των ε, γεγονότων των περασμένων μάλλον από το φως των γεγονότων των περασμένων εβδομάδων σε σχέση με το, το μεταναστευτικό και το προσφυγικό θέματα που θα πραγματευτεί κατά πάσα πιθανότητα τις επόμενες ημέρες στο Κοινοβούλιο οι βουλευτές και οι επιτροπές θα έχουν και πάλι την ευκαιρία να επανεξετάσουμε τις ε, τροπολογίε για τον προπολογισμό του 2016 με τρόπο ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις μελλοντικέ προκλήσει σε αυτό το τομέα και θα ήθελα να ακούσουμε τον κύριο Μπέγκεν με την ιδιότητα του εισηγητή να κάνει κάποια σχετικά σχόλια. Ήθελα μόνο να σας πω ότι λίγα λεπτά πριν συζήτησα με την γραμματεία και ε, οι τροπολογίες από πλευράς της Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορίου δεν μπορούν πλέον να καταταθούν διότι έχει ολοκληρωθεί σε όμως μεμονωμένοι βουλευτές μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου στις 12 μπορούν ε, να καταθέσουν άλλες τροπολογίες. Αν ένας μόνος βουλευτής ή μια ομάδα βουλευτών επιθυμούν να καταθέσουν τροπολογίες, έχουν τη δυνατότητα μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου, τις επόμενες 2-3 μέρες να το κάνουν και σίγουρα ο εισηγητής μας, ο κ. Μπέκε, θα ε, μας δώσει και περαιτέρω διευκρινήσεις. Ολοκλήρωσα τώρα τις ανακοινώσεις του Προέδρου και θα περάσουμε στο σημείο 4 παρουσίασε μελέτη σε με τίτλο Αξιολόγηση των αποφάσεων σε σχέση με την πολιτική εμπορική άμυνα για το 2014. Το 1982 έχουμε και ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ζητείται με εκπόνηση αιτήσια έκθεση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι διαδραστηριότητέ τη σε αυτό το τομέα. Τότε ήταν δύο βασικοί στόχοι. Να αυξηθεί η διαφάνεια μας επιθυμίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τόσο ώστε να λογοδοτεί για τι δράσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και δεύτερον, εξίσου σημαντικό στόχο η αιτήσια έκθεση ε, θεωρείται ένα όχημα μέσω του οποίου μπορεί να επικοινωνήσει και με το ευρύτερο κοινό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν υπήρξαν πολλά επακόλουθα ψηφίσματα μετά από αυτέ τι εκθέσει που όντω ε, συνετάξαν ετησίως και υπευλήθησαν στο Κοινοβούλιο. Για πολύ σημαντικού λόγου ε, χρησιμοποιούμε τέτοια εργαλεία για την, ε, το, την πρόταση εξυγχρονισμού των ε, μέσων της αμυντικής πολιτικής, TDI παραδείγματο χάρη. Έχουμε το θέμα του πρωτοκόλλου προσχώρησης της Κίνας στον ΟΠΟΕ με το καθεστώς της ανοιχτής οικονομίας. Για όλα αυτά τα ζητήματα είναι σημαντική η έκθεση αυτή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, το τμήμα μελετών του Κοινοβουλίου, μελέτησε την έκθεση ο κύριος Έντριν Μέλφο ε, είναι από το Πανεπιστήμιο της Βέρνης και της ε, Βαρκελόνης είναι κατέχει το ζήτημα, είναι διακεκριμένος Επιστήμος στον τομέα αυτό. Θα του δώσω το λόγο απευθείας για να μας παρουσιάσει την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στη συνέχεια θα ακούσουμε τον εισηγητή, τους συνεισηγητές και τους συντονιστές. Ο κύριος Ελμούς έχει το λόγο. Thank you very much, Mr. Winkler. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Βίνκλερ. Ίσως θα θυμίστε ορισμένοι ότι είχα εκπονήσει και μια μελέτη για την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου με θέμα το εγχείρημα εξυγχρονισμού κατά το παρελθόν, οπότε και μου είχε ζητηθεί να δώσω την προοπτική των εξαγωγιών και των εισαγωγών, αλλά και των χρηστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που μπορεί να είναι θύμα ε, κάποιων δράσεων εμπορική άμυνα για την καταπολέμηση του ντάμπινγκ. Βέβαια, όπω είναι προφανέ, άλλο είναι το περιεχόμενο αυτής της μελέτης. Ε, ανέλησα τι δύο τελευταίε ετήσιε εκθέσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπω είπε και ο κύριος Βίνκλερ όμως, ε, εγώ είμαι επαγγελματία και για να υπάρχει διαφάνεια νομίζω ότι πρέπει να γνωρίζετε ότι έχω προσωπική συμμετοχή σε πολλέ από τι υποθέσει που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εργάζομαι στο τομέα των εισαγωγών, εξαγωγών και ε, χρηστών. Το ήθελα, ήθελα να το αναφέρω για να γνωρίσετε και από πού προέρχομαι. Σε ό,τι αφορά τη μελέτη, νομίζω την είδατε, μπορείτε να τη βρείτε και στην είσοδο σε αντίτυπο. Ουσιαστικά δύο είναι τα τμήματα αυτής της μελέτης. Το πρώτο είναι μια αξιολόγηση των τελευταίων δύο ετήσιων εκθέσεων της Επιτροπής για τι δραστηριότητε της Ευρωπαϊκή Ένωσης ε, σε ό,τι αφορά την εμπορική άμυνα. Αυτό είναι το πρώτο τμήμα. Και το δεύτερο τμήμα που ε, πραγματεύομαι είναι κάποιες σημαντικές αλλαγές ε, στην αμυντική ε, πρακτική, την πρακτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι πολύ σημαντικές κάποιες από αυτές τις αλλαγές, αλλά δεν αποτελούν αντικείμενο των δύο τελευταίων ετήσιων εκθέσεων της Κομισιόν. Και αυτό δείχνει ότι οι ετήσιες εκθέσεις, ναι μεν είναι χρήσιμες σε κάποιο βαθμό, Ίσως όμως ε, να είναι και πολύ χρήσιμες για όσα δεν λέγονται και δεν συζητούνται στο πλαίσιο αυτών των ειδικών εκθέσεων. Σε το πρώτο για την αξιολόγηση δηλαδή της ετήσιας έκθεση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής εγώ εστίασα στις εκθέσεις του 12 και του 13. Για την έκθεση του 2014, ε, τη λάβαμε τον Αύγουστο, πρόσφατα λοιπόν, τον προηγούμενο μήνα. Είχε ολοκληρωθεί όμω ε, πριν ε, η μελέτη μας. Άρα καλύπτουμε τα ε, θέματα εμπορική άμυνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα έτη 2012-2013 και περιλαμβάνεται και η υπόθεση την οποία ανέφερε στην ο του κ. Βίγκλερ. Βασιζόμαστε στο ψήφισμα του 81 του Κοινοβουλίου, ένα αρκετά παλαιό ψήφισμα, που έλεγε τότε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρούσε ότι ο ρόλος του σε αυτό το τομέα είναι ότι είναι θεματοφύλακας που τα για το δημόσιο συμφέρον ε, δετάτη την ενία. Ουσιαστικά υποχρεώνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε μια αναφορά των δρασιών της και ο στόχος ε, της ε, ετήσιας αυτής έκθεσης θα είναι ένας φορέας μέσω του οποίου μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επικοινωνεί με ένα πιο πλατή κοινό. Μέχρι σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη και την τελευταία μελέτη του Αυγούστου, 33 είναι συνολικά η Εμείς αναλύουμε την 31η και την 32η έκθεση σε βάθος ε, για τα θέματα των δραστηριοτήτων εμπορικής άμυνας για το 12 και το 13 όπως είπα. Ποιε είναι οι βασικές ελλείψεις των ειδήσεων εκθέσεων. Εδώ βλέπετε μια σύνοψη βέβαια, στην έκθεση θα μπορείτε να διαβάσετε πολύ περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν σκόπιμο να συμπεριλάβω σε αυτή τη σύντομη παρουσίασή μου όλες αυτές τις ε, λεπτομέρειες. Καταρχάς, ε, τεράστια καθυστέρηση ε, μέχρι να δημοσιευθεί η έκθεση. 12 μήνες είναι η μέση καθυστέρηση των τελευταίων ετών. Ολοκληρώνεται το έτος το Δεκέμβριο, κατά μέσο όρο όμως η έκθεση θα, θα δημοσιοποιηθεί για το προηγούμενο έτος, το Δεκέμβριο του επόμενου έτους. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν εύλογοι λόγοι, γιατί είναι τυποποιημένες ε, οι εκθέσεις ουσιαστικά. Το βασικό σκορμό τη έκθεση που είναι κάποια στατιστικά στοιχεία ενημερώνονται. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θα πρέπει να δημοσιεύονται αυτές οι μελέτες, σας πάντων διατίθενται με τόσο μεγάλη καθυστέρηση. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τη μορφή της μελέτης, εγώ την αποκαλώ boilerplate, πολύ τυποποιημένη με την έννοια ότι κάθε χρόνο είναι κατά 89% ε, το ίδιο, βέβαια επικαιροποιημένα είναι τα στοιχεία και η μελέτη περιπτώσεων, η ίδια όμω είναι η μορφή, η ίδια είναι τα θέματα και σε πολύ μεγάλο βαθμό και η ανάλυση είναι ίδια κάθε χρόνο. Τρίτον, ε, υπερβολικές ή τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά μόνο σε επιλεγμένες, για επιλεγμένες υποθέσεις. Και η βάση την επιλογή αυτών των περιπτώσεων που συζητούνται στην έκθεση δεν είναι ξεκάθαρη. Με τι κριτήριο επιλέγονται δηλαδή αυτέ οι περιπτώσει. Τέταρτον, εν γέννη δεν συζητούνται ε, οι επιπτώσεις ε, που έχουν τα μέτρα σε ό,τι αφορά ε, τους στόχους τους και όταν το 1981 είδαμε ότι ο στόχος ήταν αυτός το δημόσιο συμφέρον, δεν συζητείται το δημόσιο συμφέρον τόσο πολύ σε ό,τι αφορά τα μέτρα εμπορικής άμυνας της Ένωσης. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για τις καταγγελίες ή για τις ε, ε, καταγγελίες. Σε πολλές περιπτώσεις, τα τελευταία 30 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι το 5% περίπου των ε, περιπτώσεων των καταγγελών τις ε, απορρίπτει και αυτό είναι, είναι κατά κάποιο τρόπο μια τυπική απάντηση που δίνει σχεδόν πάντοτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι εμπιστευτικά τα στοιχεία όμως, άρα κανείς δεν γνωρίζει αν αληθεύει όχι αυτό. Γιατί το λέω όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό. Το λέει για να πει ε, στο ευρύ κοινό ότι έχει υψηλά πρότυπα σε σχέση με τα σχετικά των Ηνωμένων Πολιτειών όπου προκαταβολικά ε, γίνονται πάρα πολλές ε, υποθέσεις δεκτές και μετά περατούνται πάρα πολύ γρήγορα. Ουσιαστικά γίνονται δεκτές σχεδόν όλες οι καταγγελίες. Ενώ στην πέτρηση Κομισιόν λέει το 50% αλλά με τη διαφορά ότι σε πολύ περισσότερες περιπτώσεις σχέση με τη ΣΥΠΑ έχουμε πορικά μέτρα τελικά. Καλό ε, είναι βέβαια να γίνεται καλύτερος έλεγχος εκ των προτέρων για να μην ξεκινούν ε, υποθέσεις θα πρέπει στη συνέχεια να περατωθούν ενώ δεν υπήρχε λόγος να συζητηθούν ευθύς εξ αρχής. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις, εν μέσω μιας έρευνας, Λίγη μια περίπτωση, μια υπόθεση, διότι αποσύρεται η καταγγελία. Μέσα λοιπόν στην όλη διαδικασία αποσύρεται η καταγγελία και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω σε 100% των περιπτώσεων αποφασίζει να κλείσει τη διαδικασία. Λογικό είναι αυτό βέβαια. Πρόκειται για ε, Υποθέσει του ιδιωτικού τομέα που ε, καταθέτει μια καταγγελία και αν ο ιδιωτικό τομέα αποφασίζει για οποιοδήποτε λόγο εν μέσω της έρευνας ε, να αποσύρει την καταγγελία δεν έχει λόγο να συνεχίσει την έρευνα Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαια δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο αποσύρονται οι εν λόγω καταγγελίε. Ήταν αδύναμη, ήταν, δεν ήταν πολύ ισχυρά τα στοιχεία, μήπως γιατί υπήρξε κάποιο είδου συμφωνία μεταξύ εγχώριων παραγωγών και εξαγωγή. Αυτό δεν είναι καλό βέβαια για του καταναλωτέ. αλλά όλα αυτά δεν τα αποκαλύπτουν. Ε, μόνο μία ε, σελίδα ή μισή σελίδα στην επίσημη εφημερίδα που λέει ότι αποσύρθηκε καταγγελία και θεώρησε η Κομισιόν ότι ε, καλό είναι να κλείσει αυτή η υπόθεση. Καμιά άλλη λεπτομέρεια δεν δίνεται και θεωρησε η οτι ε καλο ειναι να κλεισει αυτη κανεί που εμά δεν γνωρίζει για ποιο λόγο αποσύρονται αυτέ οι υποθέσει σε τόσε πολλέ ε, περιπτώσει. Έπειτα, δεν υπάρχει καμιά πληροφορία για τις ε, έρευνες ε, του Όλαφ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις έρευνες που είναι δαπανηρές και χρονοβόρες. Αν επιβληθούν μέτρα, γιατί βρεθεί ότι υπάρχει επιβλαβές ε, dumping, τότε τα μέτρα επιβάλλονται και πρέπει να εφαρμοστούν. Γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα, είναι αστείο, αν δεν επιβληθεί ο δασμός για παράδειγμα. Λογικό είναι λοιπόν να επιβληθούν ε, ε, τα τέλη ε, κατά του ντάμπινγκ και τα λοιπά. Αλλά αυτά θα πρέπει να εφαρμόζονται τα μέτρα και αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Στη διαδικασία με παράκαμψη μιλήσετε για τα, την υπόθεση για την Ταϊβάν και τη Μαλαισία με τα φωτοβολταϊκά και αυτές οι διαδικασίες παράκαψης δημοσιοποιούνται και είναι διαφανείς θα έλεγα. Ταυτόχρονα όμως όλα αυτά διενεργεί έρευνες στο πλαίσιο της απάτης της τελωνιακής. Παραδείγματος χάρη ψευδείς ε, δηλώσεις καταγωγής ή ταξινόμηση προϊόντων. False origin declarations τα λέμε αυτά. Δηλαδή, λένε ότι κάποιοι ότι έχουν τα φωτοβολτικά στο Χονγκ στην Ταϊβάν και δεν επιβάλλονται ε, δασμοί. Αν υπάρχουν λόγοι για την Όλαφ ε, να θεωρήσω ότι μάλλον υπάρχει απάτη, διενεργεί αυτές τις έρευνες που δεν δημοσιοποιούνται όμως ο κ. καιρών ε, κάποια ανακοινοθέντα τύπου μόνο δημοσιεύει όλα. Όμως οι έρευνε, τα αποτελέσματα των έρευνων δεν δημοσιοποιούνται σε καμία περίπτωση από την Όλαφ. Επομένω, υπάρχει ένα τεράστιο κενό ε, έλλειμμα διαφάνεια. Γιατί ουσιαστικά κανεί δεν γνωρίζει τι γίνεται από αυτή την πλευρά. Σε ό,τι αφορά τον μηχανισμό εφαρμογή ή επιβολή των μέτρων. Τέλο, τελευταία έλλειψη, αν θέλετε, τη ετήσια έκθεση είναι ότι δεν συζητούνται οι αλλαγέ ε, των πρακτικών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό είναι και το αντικείμενο του δεύτερου τμήματο τη εκθεσή μου, το οποίο θα συνεχίσω. Με το οποίο θα συνεχίσω. Ε, αλλαγέ λοιπόν στι πρακτικέ. Εμεί τι βλέπουμε ω επαγγελματίε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το γνωρίζει ότι αυτά τα θέματα δεν τα αντιμετωπίζουν οι ετήσιε εκθέσει. Δεν αναφέρονται αυτέ οι αλλαγέ. Τι έχουμε ε, παρατήρηση πρόσφατα ε, στις πρακτικές εμπορικές άμεσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ποιες είναι οι βασικές αλλαγές. Πρώτον, έχουμε πολλές έρευνες ε, για επιδοτήσεις σε σχέση με τις οικονομίες της αγοράς ξεκίνησαν το 2010. Αυτές οι έρευνες, 10 νομίζω είχαμε υποθέσεις κατά της Κίνας και πιο πρόσφατα μία κατά του Βιετνάμ. Άρα έχουμε την διενέργεια, την, ε, το άνοιγμα διαδικασιών ε, σε σχέση με τις επιδοτήσεις. Σε ό,τι αφορά αυτές τις ε, συγγνώμη, οικονομίε μία αγορά, όχι νέα αγορά. Νέε οικονομίε αγορά. Όχι, που δεν, δεν έχουν αγορά. Δεν θεωρείται αυτό δυνατό να γίνει από θεωρητική πλευρά, δηλαδή να κινηθούν διαδικασίες ε, παραβάσει για τέτοια θέματα σε χώρες που δεν έχουν ε, ουσιαστικά. Ξεκίνησε όμως αυτό ε, το 2010 περίπου ή 9 από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε αρκετές υποθέσεις τώρα. Η Κίνα είναι ο βασικός στόχος. Ένα άλλο για την Ινδία και την Κίνα για παράδειγμα, στην περίπτωση της Ινδίας, οι περισσότερες επιδοτήσεις είναι επιδοτήσεις εξαγωγών. Στις κινέζικες περιπτώσεις οι επιδοτήσεις δίνονται αν εκπληρώνονται ορισμένε προϋποθέσεις που δεν σχετίζονται με τις εξαγωγές. Δεύτερον, όπως γνωρίζετε και το είπε και ο κύριος Βίγκλερ στην εισαγωγή του, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τέλο πάντων η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποφασίσει κατά πόσο θα δώσει στην Κίνα το καθεστώς οικονομίας ε, της αγοράς ε, στα τέλη του 2016 αυτό όμως ε, μπορεί να δώσει MET σε κινέζικε επιχειρήσει, αλλά δεν γίνεται από το 11 και μετά αυτό για κινέζικες επιχειρήσεις Μάλιστα αυτό ήταν κάτι που συνέβαινε πάρα πολύ μέχρι το 11, τώρα δεν συμβαίνει. Έχουμε επίσης μια άλλη ε, τάση από το 2013 για τις προσαρμογές του κόστους ε, στους εξάγοντες παραγωγούς ε, πέραν της διπλής τιμολόγησης. Για το φυσικό αέριο τώρα και τον ηλεκτρισμό και την Κίνα ε, αυξήθηκε ε, προς τα πάνω το κόσμο παραγωγή των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ε, φυσικό αέριο και ηλεκτρισμό αυξάνεται παραγωγή και τα περιθώρια ντάμ με αυτόν τον τρόπο γιατί είναι χαμηλότερε οι τιμέ οι ντόπιε από ότι για την εξαγωγή. Από το 2013 έχει επεκταθεί αυτή η πρακτική και έχει χρησιμοποιηθεί και για τις εξαγωγές για χώρε όπως είναι το νησί και η Αργεντινή τέταρτο αυτό που κάνει από το 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι επιλέγει το δείγμα των εχώριων παραγωγών συστηματικά πριν από την έναρξη των διαδικασιών. Είναι μια συστηματική πλέον πρακτική πριν ε, ανοίξει υπόθεση. Άρα ακόμη και πριν ξεκινήσει ε, μια υπόθεση έχουν γίνει ε, κάποια ε, πράγματα και υπάρχουν και λιγότερες, λιγότερα στοιχεία τα οποία γίνονται γνωστά εκ των προτέρων. Επίσης, αυτό θα έλεγα βέβαια ότι είναι θετικό. Αυτό που έκανε και κάνει ακόμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά την επιβολή των μέτρων κατά του ντάμπινγκ, που είναι πενταετού ε, διάρκεια. Ε, τώρα η Κομισιόν ε, τα επιβάλλει για μικρότερη χρονική διάρκεια για να επανεξετάσει την υπόθεση πιο γρήγορα από ό,τι θα συνέβαινε κανονικά και η πιο πρόσφατη σχετική υπόθεση ήταν τα φωτοβολταϊκά με αποτέλεσμα του διετούς ορίου. Θα πρέπει αυτή η υπόθεση να επανεξεταστεί τα τέλη του έτου. Επίσης, τι άλλο κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε τακτά διαστήματα. Ε, ξέρει πρώτα από το πριν εφαρμογή ενό μέτρου. Δηλαδή ένα μέτρο μπορεί να καλύπτει αρχικά ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, αλλά όταν παρουσιάσουν οι ενδιαφερόμενοι ε, τις ε, του και τη ενδεχομένω ενδεχομένως ε, κάποια από τα προϊόντα που καλύπτονταν αρχικά να ε, εξαιρεθούν του πεδίου εφαρμογή όπως συμβαίνει στα φωτοβολταϊκά με ένα από τα βασικά υλικά παραγωγή όπου είχαμε κάποιες εξαιρέσεις. Επίσης, ό,τι αφορά τον υπολογισμό του περιθωρίου κέρδους, όταν υπολογίζει με βάση το lesser duty rule, τον κανόνα για το χαμηλότερο δασμό ε, της ε, ήταν σαφές από που προέρχεται ο στόχος του κέρδους. Πιο πρόσφατα, τα τελευταία χρόνια και ε, κατόπιν ε, παρότρινσης ε, του ελεκτικού συνεδρίου, η Κομισιόν έχει μια άλλη διαδικασία για τον υπολογισμό αυτού του κέρδους πριν τον Τάμπ. Και νομίζω ότι μπορώ εδώ να ολοκληρώσω την παρουσίαση. Με ευχαριστώ. Uh, uh, ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Κοιτάξτε, προφανώς δεν έχω το κύρος της Επιτροπής του κύριου Λάγκε, ο οποίος ε, χρησιμοποιεί ε, αυτό το σφυράκι, αλλά θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει αυτή η ομιλία, έχει διανομηθεί, ποιος θέλει λοιπόν μπορεί να μπει σε λεπτομέρειες. Θα ήθελα λοιπόν επίσης ε, πριν ξεκινήσει η συζήτηση για αυτό το σημείο της μέρης διάταξης, να σας πω ότι και στο επόμενο σημείο θα συζητήσουμε για το ίδιο θέμα και θα έχουμε και συζήτηση με την Κομισιόν και κλεισμένων των θυρών. Ας περιοριστούμε λοιπόν τώρα σε αυτή τη μελέτη και αργότερα θα αναφερθούμε στο ίδιο θέμα, αλλά από κοινό ε, με την Κομισιόν. Ο κύριος Φιέντλ θα λάβει το λόγο. Ήταν ε, ο εισηγητής ε, της, του TDI, ο Κρίστοφερ έχει το λόγο. Κοιτάξτε, περιμένουμε ακόμα το Συμβούλιο να μας υποβάλει την πρότασή του και μέχρι τότε εγώ εξακολουθώ να παραμένω εισηγητής. Μπας περιπτώσει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη μελέτη σας. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, το θέμα των ερευνών της Όλαφ. Εξηγήσατε βέβαια κάποια πράγματα, αλλά από ό,τι θυμάμαι ε, είχαμε τον πρώην ε, τμήματάρχητο επικεφαλής ε, της Όλαφ, ο οποίος είχε υποσχεθεί να εξετάσει συγκεκριμένα μέτρα TDI. Τώρα, όσον αφορά την ε, μεταχείριση της οικονομίας της ε, αγοράς. Στο κείμενό σας υπάρχουν κάποιες εξηγήσει, αλλά διερωτώ με, κατάλαβα καλά ότι αυτό είναι κάτι ε, το οποίο προκαλεί σοβαρές ανησυχίες και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γιατί αν θυμάμαι καλά, τουλάχιστον τρεις φορές η άρνηση της Κομισιόν να δεχτεί ε, και να δώσει κάποιες επιχειρήσεις τη μεταχείριση οικονομίας της αγοράς, αυτό το έχει αμφισβητήσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τρίτον, ασκήσατε κριτική όσον αφορά στη διαφάνεια. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας ε, ερωτήσω αν μπορείτε να μας πείτε λιγάκι ποια είναι η διαφορά εδώ στην Ευρώπη σε σχέση με την Αμερική. Γιατί αν θυμάμαι καλά εκεί χρησιμοποιούν για το EPO στην Αμερική και αυτή η δυνατότητα ε, επιτρέπει στους δικηγόρους ε, να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στη διαφάνεια. Βέβαια, ο κίνδυνος είναι ότι αν διαρρεύσουν στοιχεία μπορεί να αποκλειστούν από το δικηγορικό σύλλογο. Πιστεύετε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να γίνει το ίδιο. Και τέλος, να ρωτήσω το εξής. Είπατε ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για την απόσυρση καταγγελιών. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι η Κομισιόν γνωρίζει τα αίτια της απόσυρσης καταγγελιών. Ε, εντάξει, μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι ενδεχομένως δεν διαπίστωσε ζημιά, αλλά ε, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα έγγραφα όπου μια εταιρεία ε, να λέει με έγγραφο ότι αποσύρουμε την καταγγελία και αφού δεν γίνεται αυτό τότε οι κατάλογοι αυτοί της Κομισιόν δεν είναι περισσότερο. Οι κασίες υποθέτουν δηλαδή ότι έγιναν αυτές οι αποσύρσεις καταγγελιών. Αυτές είναι οι τρεις ερωτήσεις που είχα να υποβάλω. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ Κρίστοφα. Και τώρα ε, οι συντονιστές, αν επιτιμούν, ε, μπορούν να λάβουν το λόγο με την συνήθη σειρά. Αν βέβαια δεν επιτιμούν οι συντονιστές το λόγο, κατόπιν τα μέλη της Επιτροπής μπορούν να λάβουν το λόγο. Η Αλέξια Μόσκα. Κοιτάξτε, εγώ έχω να κάνω αρκετές ερωτήσεις, κυρίως ε, όσον αφορά ε, στην άποψη της Επιτροπής γιατί με ενδιαφέρει να ενημερωθώ περισσότερο για το με βάση αυτή τη μελέτη, τι είδους δράσεις μπορούν να λάβουν χώρα. Εγώ λοιπόν θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις στο δεύτερο σκέλος της μελέτης. Βέβαια και εγώ θα ήθελα να έχω ή δυνατόν κάποιες περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όλα αυτά που αναφέρθηκαν. Κοιτάξτε, από τη μία έχουμε τις αλλαγές ε, οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε επίπεδο Ηνωμένων Πολιτειών. Όσον αφορά δηλαδή τα δικά τους εργαλεία για την ε, εμπορική άμυνα. Και θα θέλαμε να ξέρουμε αυτές οι αλλαγές γιατί προέκυψαν, για ποιο λόγο και πώς είναι δυνατόν να διαπιστώσει κανείς ε, αν υπάρχει ομοιογένεια στη μεταχείριση. Αυτό είναι το ένα. Και από την άλλη πρέπει να πω ότι είναι μια ερώτηση που αφορά βέβαια περισσότερο αργότερα τη συζήτηση που θα ακολουθήσει με την Κομισιόν, αλλά θα το ρωτήσω τώρα. Λοιπόν, με βάση τις ε, αλλαγές που αυτή τη στιγμή έχουν μπλοκαριστεί στο Συμβούλιο και εκεί δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ξεμπλοκάρισμα της όλης κατάστασης, εγώ διαρωτώ με. Ποιες αλλαγές ε, συμβαδίζουν με τις ε, αλλαγές και είναι σωστό ότι σήμερα έχουμε προχωρήσει ένα βήμα πιο κάτω στη διαφάνεια. Και βεβαίω ε, μετά που θα στήσουμε με την Επιτροπή θα τα ξαναπώ αυτά, αλλά να πω και τώρα ότι κατά την άποψή μου τα βήματα εμπρό στον τομέα της διαφάνειας που έλαβαν χώρα δεν αρκούν γιατί για μας, ε, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει και εμείς ε, να μπορούμε να ελέγχουμε, να ελέγχουμε το κατά πόσον είναι δυνατόν να υπάρξει κάποια βελτίωση στο θέμα της διαφάνειας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Σόλτς έχει το λόγο. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω για τη συζήτηση σχετικά όμως που αυτή η συζήτηση μάλλον είναι του 5 όχι του 4, είναι του σημείου 5 της μέσης διάταξης, αφορά περισσότερο τη συζήτηση με την Κομισιόν. Αν κατάλαβα λοιπόν καλά, εσείς είπατε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο του, του θεματοφύλακα των εμπορικών πολιτικών και αυτό λόγω των πληροφοριών που αποκτούμε κάθε χρόνο από την έκθεση Κομισιόν. Και ρωτώ, αν είναι έτσι τα πράγματα, τότε τι έχετε να μας συστήσετε σε αυτή την Επιτροπή και γενικότερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Κρίστοφε είπε ότι περιμένει ακόμα την άποψη του Συμβουλίου, άρα όλοι περιμένουμε. Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση είναι η εξής με ενδιαφέρει να γνωρίζω την προσέγγιση άλλων κρατών σχετικά με τα δικά τους τα εργαλεία εμπορικής άμυνας, Trade Defense Instruments. Το θέμα δεν είναι αν θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερο εμπόριο ή προστασία. Ε, το θέμα που δείτε είναι ο εμπορικός πόλεμος. Ποια είναι τα στοιχεία που αφορούν σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες χώρες και επίσης στο πλαίσιο του ΠΟΕ πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε γενικότερα μια πολιτική εξυγχρονισμού των ε, εμπορικών αυτών πρωτοβουλειών. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος επιθυμεί να λάβει το λόγο. Αν όχι, θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή δεν ξέρω αν η Επιτροπή θέλει τώρα να παρέμβει σε σχέση με τη μελέτη. Επιτροπή θέλετε να λάβετε το λόγο. Κύριε Γουίνκλερ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα κι εγώ επί τη ευκαιρία να κάνω κάποιες παρατηρήσεις ο πλευρός του κυρίου Φάλμεστη. Πρώτα απ' όλα είναι ξεκάθαρο για μας με την περιγραφή που γίνεται μέσα στην έκθεση για τις ε, λήψεις και τις ατέλειες ότι ε, εσταθούν αυτά τα στοιχεία, δεν αμφισβητεί κανείς ε, την κατάσταση όπως την περιγράφει ο κύριος Γουίνκλερ. Ε, τούτο έχουμε κάποιο ζήτημα με τις συστάσεις μέσα στην έκθεση και θα ήθελα να σχολιάσω τις παρατηρήσεις αυτές κύριε Γουίνκλερ χοντρικά λέει η έκθεση να μας δίνετε τις εκθέσεις μέσα σε τρεις μήνες, αλλά διπλάσεις, δηλαδή θέλουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Από τη δική μας οπτική γωνία δεν συνάδουν αυτά τα δύο και δεν σημαδίζουν αυτά τα δύο και δεν συνάδουν και με την, το στόχο της έκθεσης ο οποίος είναι να κάνει μια επισκόπηση και όχι μια απογραφή όλων των σχετικών δράσεων ε, ε, αμυντικής εμπορικής πολιτικής, ε, διότι έχουμε και άλλα μέσα στη διάθεσή μας που είναι και προσβάσιμα. Οι εκκρεμείς υποθέσεις είναι όλες στον ιστότοπό μας. Η αποφάση του δικαστηρίου είναι στον ιστότοπο του δικαστηρίου. Επίσης, ε, όσοι κάνουν τις ακροάσεις έχουν εκθέσεις δραστηριότητες και αυτά είναι διαθέσιμα, αλλά ξεχωριστά. Υπάρχουν όλα αυτά. Το 82 δεν υπήρχαν, αλλά τώρα όμως υπάρχουν και δεν επιθυμούμε να υπάρξει επικάλυψη των προσπαθειών. Για την Όλαφ μπορώ να σας πω ότι σε κάποιες ε, από τις έρευνες, κυρίως για την παράκαμψη των μέσων ε, εμπορικής πολιτικής, ε, ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα. Δηλαδή, οι αρχές των τρίτων χωρών, των χωρών που συνεργάζονται μεταξύ μας, ε, τηρούν αυτήν την αρχή της εχεμήθειας, ούτως ώστε να μπορέσουν να συλληφθούν αυτοί που κάνουν τις πλαστές δηλώσεις. Σχετικά τώρα με τον χρόνο υποβολή τη έκθεση, όντω θα μπορούσε να γίνει και συντομότερα. Ε, εμείς θα καταφέρουμε μέσα σε 6 μήνες, γιατί ο μέσο είναι 12 μήνες, ε, και κατέστη διαθέσιμη η έκθεση τον Αύγουστο, μπορούμε βεβαίως να κάνουμε μεγαλύτερες προσπάθειες και να την έχουμε έτοιμη το Πάσχα. Όταν ε, σε σχέση με το καθεστώς ε, οικονομίας της αγοράς υπάρχουν σοβαρές εξελίξεις, ε, μπορούμε να είμαστε και πιο και πιο, να υποβάλουμε πιο περιστατωμένες εκθέσεις και να αιτιολογούμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια για τις επιλογές που κάνουμε, που κάνουμε μέσα στην έκθεσή μας για τα μέτρα που πρέπει να αναλυθούν. Ε, νομίζω ότι ήταν χρήσιμες παρατηρήσεις, κύριε Φελμούς. Για τα εμπορικά ζητήματα, φυσικά αξίζει να συζητήσουμε, αλλά μπορούμε να ε, αντιστρέψουμε την ερώτηση και να σας υποβάλουμε ακριβώ την ίδια ερώτηση γιατί ε, αυτά τα ζητήματα. Εσείς μας είπατε γιατί διαλέξατε αυτά τα πέντε, σας ρωτούμε και εμείς γιατί διαλέξατε εσείς αυτούς τους πέντε τομείς σα διαβεβαιώ ότι δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση πολιτική μεθόδευση. Δηλαδή, ε, είπε κάποιο το 2011 ότι δεν μπορεί πλέον να χορηγηθεί καθεστώ ε, αρχή ε, οικονομία τη αγορά. Ε, λοιπόν, εξετάζεται η υπόθεση από το δικαστήριο, γίνεται αναθεώρηση και αν δεν είμαστε ικανοποιημένοι ότι υπάρχει μόρφωση με τα πέντε κριτήρια, οφείλουμε να απορρίψουμε την αίτηση. Για τι ε, υποθέσει, ε, για τι επιδοτήσει, όντω το κάνουμε και αυτό σε σχέση με το καθεστώ οικονομία τη αγορά ε, και προσφάτως έχουμε χρησιμοποιήσει και αυτή τη μεθοδολογία σε μια περίπτωση διπλής τιμολόγησης και εκκρεμεί η υπόθεση στη Γενέβη. Ε, η Αργεντινή είχε κάνει την προσφυγή και θα συμφωνήσω και με τον διακεκριμένο εμπειρογνώμων ότι ε, στην φάση προδρομολόγησης δεν είμαστε σίγουροι ότι βελτιστοποιείται η διαδικασία όταν ε, προσέρχονται τα μέρη και ανταλλάσσουν ε, δειγματοληπτικά στοιχεία. Ε, διότι για μια πενταετή περίοδο ίσως χρειάζεται περιορισμός του καταλόγου των αγαθών. Γενικά θα έλεγα πως με τους περιορισμούς ε, της νομοθετικής ε, ρύθμισης ε, πληρούμε το ρόλο μας για, την, για το δικαστικό έλεγχο των υποθέσεων. Σας ευχαριστούμε και τώρα θα ακούσουμε τον Δόκτωρο Φελμούστο. Είναι μάλλον πρόκληση το να απαντήσετε, αλλά παρόλα αυτά σας παρακαλώ να περιοριστείτε στα 5 λεπτά, διότι είναι πολύ φορτωμένη η ημερήσια διάταξη. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αρχίζω με αυτά, τις παρατηρήσεις του κυρίου Φιέλνα. ότι το καθεστώς, ε, η, η άρνηση του καθεστώτος χορήγης, της χορήγης του καθεστώτος της οικονομίας της αγοράς ε, είναι ένα ε, δεδομένο και μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν προσφυγές στο δικαστήριο, όμως ε, το γεγονός είναι ε, Κανένα δεν πήρε τέτοιο καθεστώ εμήθη σε περίπτωση επιστροφή και διάφορε τέτοιε υποθέσει εκκρεμούν. Δηλαδή, επιχειρήσει που έχουν λάβει αυτό το καθεστώ, αλλά ε, ε, μετά υπήρξε ανάκληση του καθεστώτο. Ε, χρειάζονται 5-6 χρόνια εξάλλου για τη διεκπαιρέωση αυτών των δικαστικών υποθέσεων, αλλά δίκιο έχετε κύριε Φιέλνερ ότι έχει κατατεθεί έφεση. Για την απόσυρση, την ανάκληση, Μπορούμε ίσω να το εξηγήσουμε και στην επόμενη συνεδρίαση που γίνεται για κλεισμό των ε, σειρών, αλλά μπορώ να σα πω ότι ε, είμαι 99% σίγουρο ότι στο 100% των περιπτώσεων ξέρει πολύ καλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί ε, προτάσει αυτή την άρνηση, διότι γίνεται ένα έλεγχο. Δεν είναι ότι πάτε και λέτε Α, αυτή είναι η άποψή μου και παρακαλώ να την δεχτείτε. Όχι. Γίνεται πολύ εμπεριστατωμένη ανάλυση από πλευρά των υπηρεσιών τη Ευρωπαϊκή επιτροπή, Δηλαδή δεν μπορεί να κάποιος απλώς να πάει «Α, ε, έχω αποσύρει τώρα, θα επιθυμώ να αποσύρω την υποθέση μου, ξεχάσετε τι κι εσεί. Δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει επιχειρηματολογία, υπάρχει αιτιολόγηση για την απόσυρση μια υπόθεση, μιας προσφυγής που έχει κατατεθεί. Επίσης, για το θέμα της διαφάνειας, ε, όπως προκύπτει από την έκθεση, υπάρχει ένα πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το πρόβλημα δεν είναι το, το κανόνας του lesser duty. Ε, έχουμε τις, τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως εξακολουθεί να υπάρχει ένα πρόβλημα διαφάνειας όπως το σύστημα EPO, το ΙΠΑ, που βελτιώνει ε, σαφέστατα ε, την κατάσταση ως προς τη διαφάνεια. Αυτό μας λέει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Μόσκο, κύριο Σόλτς τώρα, με ρωτήσατε τι γίνεται στη ΣΥΠΑ για κάποια από αυτά τα ζητήματα. Δεν υπάρχει τέλειο σύστημα. Έχουμε και εμείς καλά δυνατά σημαία και αντίθετα έχουν και οι ΕΠΑ. Θα συμφωνήσουν νομίζω όλοι όμως ότι είναι κατά πολύ διαφανέστερο το αμερικανικό σύστημα. Όλοι ξέρουν τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια ε, διεκπαιρέωση μιας υπόθεσης. Ε, οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, όμως ε, το αποτέλεσμα είναι χειρότερο σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό ισχύει και για τους ε, δασμούς αλλά και για τις επιδοτήσεις. δηλαδή το αποτέλεσμα είναι χειρότερο, όμως η διαδικασία είναι κατά πολύ διαφανέστερη. Λοιπόν, εγώ εκεί εντοπίζω τη βασική διαφορά ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι το πρόβλημα ότι πολλοί αντιγράφουν το σύστημα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρε όπω η Ινδία, η Κίνα, η Βραζιλία, το Μεξικό εμπνέονται και αντιγράφουν το σύστημα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι τα καλά του σημεία. Ε, αλλά κάρτε επιλέγουν αυτά τα σημεία που τους ενδιαφέρουν και για τη διαφάνεια δυστυχώ ακολουθούν το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Σμόλς, μας ρωτήσατε για, την, ε, για τα θέματα εξυγχρονισμού. Νομίζω αυτό είναι θέμα ε, που πρέπει να συζητηθεί και κλεισμένο των θύρων. Μάλλον δεν έχω να σα δώσω συγκεκριμένη απάντηση. Στη μελέτη που έχω κάνει πριν από δύο χρόνια έχω δώσει κάποια στοιχεία. Νομίζω ότι η Επιτροπή ΙΝΤΑ Διεθνού Εμπορίου δηλαδή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπερβάλλει σε σχέση με, την, ε, με τις σε σχέση με τη μεταρρύθμιση της πρότασης Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και γι' αυτό έχει δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση στα κράτη-μέλη. Δεν μπορώ να σα πω περισσότερα. Ο κ. Χόφμαν ε, έκανε πολλέ παρατηρήσει. Ένα μόνο θέλω να σχολιάσω. Με ρωτήσατε γιατί εγώ επέλεξα αυτή τα 7 σημεία, ε, δηλαδή σημαντικές αλλαγές στις πρακτικές Ευρωπαϊκές Επιτροπές. Ε, μα γιατί από τη δική μου πλευρά αυτά ε, έχουν τη μεγαλύτερη βαρύτητα αν λάβει κανεί υπόψη τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια. Αν εσείς έχετε να προσθέσετε και κάτι άλλο, πολύ ευχαρίστω να το συμπληρώσω στην επόμενη εκδοχή της έκθεσής μου. Αυτά, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε εδώ πέρα, και τώρα θα στραφώ προς τον εισηγητή μας αν χρειάζεται να κάνετε κι εσείς κάποιες παρατηρήσεις κύριε Φιέλνερ. Ευχαριστώ. Τίποτα δεν έχω να προσθέσω. Καλά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση και ολοκληρώνεται τώρα η συζήτηση για αυτό το σημείο αλλά και για το θέμα, διότι θα συνεχίσουμε για το ίδιο θέμα Θα αρχίσει η κεκλεισμένο των θυρών συνεδρίαση τώρα και παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, η Βοηθή τους, η Νομική Υπηρεσία, οι υπηρεσίες, οι υπάλληλοι συγγνώμη των πολιτικών ομάδων να παραμείνουν και όλοι οι υπόλοιποι ε, να αποχωρήσουν, παρακολούνται. Και, ε, θα παρακαλούσαμε να γίνει σύντομα, διότι δεν έχουμε χρόνο στη διάθεσή μα. Η χρονοθυρίδα που έχει προβλεφθεί για διακλεισμό των θηρών συνεδρίων είναι 35 λεπτά.